So, dear colleagues, may we begin? Αξιότιμοι συνάδελφοι, παρακαλώ πάρτε θέση να ξεκινήσουμε. Uh, do you hear me? Με ακούτε? Do you hear me now? Τώρα με ακούτε? And now you, do you hear me now? Με ακούτε? Πολύ ωραία, έτσι φαίνεται. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έγκριση τη μίληση διάταξη. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να σα ενημερώσω για, τα, για τι εξή αλλαγέ στο σχέδιο μίληση διάταξη. Στα σημεία 4, 1. 14, 15 και 18 αναβάλλονται. Το 6 θα εξεταστεί μετά το 12. Το σημείο 14 επίσης θα εξεταστεί μετά το 22. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις αυτές τις αλλαγές στην μεσοδιάταξη, οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται. Και τώρα ανακοινώσει του Προέδρου. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις αποφάσεις των συντονιστών. Στη συνεδρία σήμερα το απόγευμα, οι συντονιστές πήραν τις εξής αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα να επαληθεύσουν επί τη βάση του κανόνα 39 την καταλληλότητα της νομικής βάσης όπως αυτή αναφέρεται στην προσωρινή συμφωνία μεταξύ των συνομοθετών ε, που επετεύχθη στις 12 Φεβρουαρίου για την ευθυγράμμιση του RPS στην πρόταση Omnibus. Εάν χρειαστεί τώρα και στην περίπτωση που η προσωρινή συμφωνία μεταξύ των συνομοθετών επιτευχθεί για τους whistleblowers, να επαληθεύσουμε ότι με βάση του κανόνα 39.3 είναι κατάλληλη νομική βάση που προβλέπεται σε αυτή την προσωρινή συμφωνία. Τρίτον, να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει και να συζητήσει στην Επιτροπή μας την, ε, το νέο σημείο από του φορεί για την απόσυρση του Βασιλείου ε, και του κανόνες τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της, ε, του αστικού δικαίου και του διεθνούς, ιδιωτικού δικαίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την δημόσια ακρόαση ανάκτηση ε, οφειλών, αυτή αναβλήθηκε. θα γίνει κάποια στιγμή στο πρώτο εξάμεινο του 2019. Επίσης θα καλέσουμε έναν εκπρόσωπο της ομάδας ψηλού επίπεδου για το μέλλον, ε, σε μια μελλοντική συνεδρίαση μάλλον, ε, για το θέμα της ε, τεχνητής δεν ξέρουμε πότε ακριβώς, και τέλος θα πρέπει να γίνει μια ψηφοφορία για την προσωρινή συμφωνία που προέκυψε από τις διαθεσμικές διαπραγματεύσεις ε, για το copyright ε, στην ψηφιακή αγορά. Αυτό θα γίνει σε μια εξαιρετική συνεδρίαση ε, έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας για τον φάκελο SPC στις 26 Φεβρουαρίου πιθανότατα στις 3 αυτά για τις ανακοινώσεις και τώρα συνεχίζουμε με την ψηφοφορία ελπίζω να έχετε όλοι την κάρτα ψηφοφορίας, να την έχετε έτοιμη. Ξεκινούμε λοιπόν Uh, λοιπόν, σημείο 4.2 άσυλο και μετανάστευση, ταμείο ασύλου και μετανάστευσης. Πριν ψηφίσουμε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Λεμπρετών εάν δεν έχετε αντίρρηση. Εάν το επιθυμεί βέβαια ο ίδιος. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα πολύ σύντομα να πω δύο λόγια το αντικείμενο αυτής της πρότασης είναι η δημιουργία ενός ε, ταμείου ασύλου και μετανάστευσης που θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. Ε, έχει ως στόχο την ε, διαχείριση των μεταναστευτικών ορών. Δεν θα μιλήσω τώρα επί της ουσίας, διότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ένα πρόβλημα νομικής βάσης εδώ. Είναι προφανές ότι τα άρθρα 78 και 79 της συνθήκης είναι τα κατάλληλα άρθρα, μιας και σχετίζονται με την κοινή πολιτική μετανάστευσης, Όμω υπάρχουν αμφιβολίε για το άρθρο 80. Μια και το άρθρο 80 είναι πολύ γενικό, αναφέρεται σε μια αρχή αλληλεγγύης, στην ισότιμη κατανομή των ε, ευθυνών ε, μεταξύ κρατών μελών και σε οικονομικό επίπεδο όπου αυτό χρειαστεί. Πολύ λοιπόν ασαφές το άρθρο αυτό και δεν είμαι πεπισμένος ότι είναι κατάλληλο ε, για αυτή τη νομική βάση. Πρώτα απ' όλα Πρόκειται για ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται ουσιαστικά σε ένα πολύ ευρύ στόχο, πολύ γενικό στόχο. Είναι πολύ ασαφέ για να αποτελέσει νομική βάση, δεν έχει να προσθέσει κάτι στα άλλα άρθρα, το 78 και το 79. Επίση, ε, εάν θέλουμε να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για νομική βάση διακριτή, ε, νομίζω ότι αυτό αντιβαίνει την ομολογία του δικαστηρίου. Ιδιαίτερα στην απόθεση σε 411 του 2009 που υπενθυμίζει ότι οι πολλαπλές νομικές βάσεις μπορεί να γίνουν αποδεκτές μόνο όταν έχει πολλαπλούς στόχους το νομοθέτημα. Πολλαπλούς στόχους ίσης σημασίας, ενώ εδώ ο στόχος είναι ένας. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτή τη σύσταση, να αποφύγουμε τις πολλαπλές νομικές βάσεις. Και τελευταίο στοιχείο, όταν ο κανονισμός ε, για το προηγούμενο ταμείο είχε εγκριθεί, τότε δεν υπήρχε καμία αναφορά στο άρθρο 80. Υπάρχει δηλαδή και προηγούμενο εδώ. Ε, αυτή η επιλογή μάλιστα έγινε μετά από συζήτηση. Είχε γίνει μια συζήτηση για το κατά πόσο θα έπρεπε να προσταθεί το άρθρο 80 στη νομική βάση και τότε αποφασίσαμε να μην το κάνουμε. Οπότε, όπως βλέπετε, εδώ έχουμε μια σειρά από επιχειρήματα. Για να είμαι όμω πλήρη, από την άλλη, υπάρχει ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου με ημερομηνία 26 Μαρτίου 2016 για την κατάσταση στη Μεσόγειο, που διατύπωσε την επιθυμία να προσθεθεί το άρθρο 80 στα άρθρα 78 και 79. Βεβαίως αυτό είναι απλά μια επιθυμία, μια ευχή. Η νομική βάση είναι κάτι το, οποίο δεν μπορούμε να, το, να την προσθέτουμε κατά το δοκούν. Τώρα, ε, συνοψίζοντας, για το 78-79 δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, για το κατά πόσο θα πρέπει να προσθεθεί και το άρθρο 80 στην νομική βάση, εγώ ε, προτείνω να καταψηφίσουμε μια τέτοια επιλογή, να ακούσουμε και την άποψη τη νομική υπηρεσία ενδεχομένω για το ζήτημα. Θέλετε το λόγο, κυρία αλλά ναι, παρακαλώ. Ναι, δεν είμαι πολύ σίγουρη για αυτά που λέει ο κ. Λεμπρετόν. Εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει να συζητήσουμε κατά πόσο πρέπει να προσθεθεί μια νομική βάση σε αυτή την πρόταση ή όχι. Εμεί είμαστε υπέρ. Δεν μιλάμε εδώ για την πρόταση και τη γνώμη του εισηγητή. Να μας εξηγήσει όμως η νομική υπηρεσία, κακό δεν κάνει. Η νομική υπηρεσία θέλει το λόγο, Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσουμε τι είναι μια νομική βάση. Η νομική βάση είναι μια διάταξη, ένα άρθρο της συνθήκης που δίνει τη δυνατότητα στα θεσμικά όργανα να πάρουν μια απόφαση. Αυτό. Τόσο απλό. Τι σημαίνει αυτό. Είναι πάντα μια διάταξη της συνθήκης λοιπόν που προβλέπει μια διαδικασία λήψης αποφάσεων. Βλέπω λοιπόν το άρθρο 80. Το άρθρο 80 ε, δεν ανταποκρίνεται σε κάποια λήψη απόφασης. Το άρθρο 80 ορίζει έναν στόχο. Έναν στόχο που έρχεται να προσθεθεί στους επιμέρους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 77, 78 και 79 και που έχουν να κάνουν με τη διέλευση των συνόρων, το άσυλο, και τη μετανάστευση. Γι' αυτό υπάρχει ένα άλλο άρθρο, το άρθρο 80, διότι η αρχή της αλληλεγγύης ισχύει και εφαρμόζεται και για τα τρία προηγούμενα άρθρα. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι το άρθρο 80 δεν είναι από μόνο του μία νομική βάση. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την ιδέα στην πρόταση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ να προσθεθεί αυτό το άρθρο στη νομική βάση, αυτό δεν θα έχει κάποιες νομικές επιπτώσεις αρνητικές. Δεν αλλάζει κάτι στην πραγματικότητα. Αυτό που θα συμβεί πιθανότατα είναι ότι όταν θα πρέπει να συντάξουμε την νομοθετική πράξη και η νομική από διάφορα θεσμικά όργανα θα χρησιμοποιήσουν το μοντέλο των νομοθετικών πράξεων ε, της Ένωσης θα δούμε ότι μόνο αυτές οι νομικές βάσεις μπορούν να συμπεριληφθούν και το άρθρο 80 ε, σίγουρα ε, μπορεί να αναφέρεται ε, κάπου αλλά όχι στο διατακτικό της νομοθετικής πράξης. Βεβαίως ε, το περιεχόμενο της νομοθετικής πράξης αναφέρεται στην νομοθεσία και δεν υπάρχει πρόβλημα αλλά δεν αποτελεί νομική βάση. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ακούσαμε την πρόταση του εισηγητή να μην προσθεθεί το άρθρο 80 της συνθήκης Λοιπόν, να προσέξουμε τι ψηφίζουμε, έτσι. Ποιος Οποιο δεν θέλει το άρθρο 80 ψηφίζει υπέρ, έτσι. Όποιος θέλει να φύγει το άρθρο 80 θέλει, ψηφίζει υπέρ. Οποιο θέλει το άρθρο 80 ψηφίζει κατά της πρόταση του εισηγητή, έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. It has been rejected. Απορρίφθηκε. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπέρ του άρθρου 80 και της συμπερίληψής του. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο 4-3. για την ετοιμότητα ε, σε περίπτωση κινδύνου στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Κύριε Λεμπρετών, θέλετε το λόγο και πάλι. Ναι, πολύ σύντομα, εδώ δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πρόκειται για μια πρόταση κανονισμού που θεσπίζει κοινού κανόνες για την διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την διαχείριση και την πρόληψη των κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Προτείνεται το άρθρο 194 παράγραφος 2 νομική βάση που είναι η κατάλληλη νομική βάση, μιας και το άρθρο αυτό αναφέρεται στην ενέργεια, στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης. Σωστό λοιπόν το άρθρο αυτό. Μάλιστα, ακούσατε λοιπόν την πρόταση, άρχιτη ψηφοφορία. And it has Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Λεμπρετό. Και συνεχίζουμε. Τώρα και κλεισμένο το θυρών. Θα ήθελα να ρωτήσω όλους όσους ε, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση αυτή ε, και το των θυρών να αποχωρήσουν.